πρόεδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνουμε την ε, συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ενημερώσω ότι τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν ήδη διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στις δηλώσεις του συμβουλίου και